της οδηγίας της σχετικής με τους ιστούς και τα κύτταρα. Ευχαριστώ Επίτροπε. Θα ήθελα να πω ότι η συζήτηση τελείωσε και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις, 10, ε, στις 12. Συγγνώμη. Και τώρα κυρίες και κύριοι πάμε στο επόμενο θέμα της μελισσίας διάταξης που προβλέπει την έκθεση του κυρίου Γκούσταυσον για το ρόλο των γυναικών στην πράσινη οικονομία. Ο κύριος Γκούσταυσον έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Από την πρώτη κιόλας μέρα και κατά τη διάρκεια στη συνέχεια της ε, εργασίας μου συνολικά Είχα πάντα καλή συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές με τους συνεργάτες διαφορετικών οργανώσεων. Θα ήθελα τις πιο θερμές μου ευχαριστίες να απευθύνω σε όλους εκείνους που συνεργάστηκαν και συνεισέφεραν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Οι απόψεις τους συνεισέφεραν στο να είναι μια ε, σφαιρική παρουσίαση απόψεων είτε μέσω τροπολογιών είτε μέσω προφορικών παρεμβάσεων και παρατηρήσεων Συμπεριλήφθηκαν πολλές λοιπόν διαφορετικές απόψεις. Πρόκειται για μια σφαιρική υπερκομματική έκθεση όπου διαφορετικές ε, παρεμβάσεις ε, συγχωνεύονται και συγκλίνουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ιδιαίτερα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσεως. Πρόκειται για οικονομικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οι λύσεις ε, και επιλύσεις αυτών των οικονομικών προβλημάτων πολλές φορές διαμορφώνονται με πολύ τεχνικό τρόπο τόσο τεχνικό λες και δεν θα υπήρχε άλλη δυνατότητα να δράσει κανείς. Ιδιαίτερα όταν έχουμε έναν πλανήτη του οποίου οι πόροι είναι περιορισμένοι, είναι πεπερασμένοι και το σημερινό σύστημα δεν λαμβάνει φυσικά υπόψη το πεπερασμένο των φυσικών πόρων, του φυσικού πλούτου. Η διαρκής ανάπτυξη έχει ε, μια συνιστόσα θρησκευτική θα έλεγα στην αιμονή με την οποία ακολουθείται και εφαρμόζεται. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πόροι, οι υδάτινοι πόροι, το νερό, η ενέργεια, ε, τα ορυκτά, τα μέταλλα, όλα αυτά έχουν επιπτώσεις ε, στους ίδιους τους φυσικούς πόρους. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ισορροπημένη πράσινη οικονομία, μια αηφόρο οικονομία πράσινου χαρακτήρα που θα έχει την αηφορία ως στόχο της και την ισορροπία που θα προσπαθεί να διασφαλίσει λαμβάνοντας υπόψη και τις ανθρώπινες ανάγκες. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι θα υπάρχει μια ισοδίκαιη δίκαια κατανομή των πόρων σε σχέση με τους κατοίκους ε, της οικουμένης. Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών επίσης. Η πράσινη οικονομία δεν είναι μόνο η πράσινη τεχνολογία, είναι και η κοινωνική δικαιοσύνη Πρόκειται για ένα ευρύτερο πλαίσιο αηφορία το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε και να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τις αγορές και τους βραχυπρόθεσμους ε, στόχους σε σχέση με τις αγορές αλλά σε ένα πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο να σεβόμαστε τις επιθυμίες των ανθρώπων, των πολιτών και να υπάρχει η αηφορία, η οικολογική αηφορία. Η οδός πρέπει να ε, στοχεύει στην πράσινη οικονομία, στο πρασινό σύνισμα της οικονομίας, στην οικολογική δράση. Πρέπει η αηφορία να εντάσσεται στην, στα πρότυπα κατανάλωσής μας και στα πρότυπα δράσης μας. Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, καταναλώνουμε και εκμεταλλευόμαστε τους πόρους, ε, τους φυσικούς πόρους, με, με άνισο τρόπο και όσον αφορά τους πόρους, αλλά και με άνισο τρόπο σε σχέση με άνδρες και γυναίκες. Πρέπει να πάψει να ισχύει αυτό το πρότυπο και να υπάρχει υπάρχει η δικαιοσύνη η οποία θα εισαχθεί. Στις μεταφορές για παράδειγμα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα στοιχεία φορεία. Είναι όλοι αυτοί συναφείς τομή, ε, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαφορετικότητα των προτάσεών μας. Μια ολόκληρη σειρά προτάσεων που θα οδηγήσουν σε μια αηφόρο οικονομία όπου άνδρες και γυναίκες από κοινού θα καθορίζουν και θα προσδιορίζουν τη μελλοντική ανάπτυξη και τα οικοσυστήματα της οικουμένης θα μπορέσουν να διασφαλιστούν και να διατηρηθούν. Ευχαριστώ. Ξεκινούμε τη διαδικασία Catch the Eye. Τώρα στη συνέχεια η κυρία Ζαμπόσκα, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ. Θα ήθελα συνοπτικά να αναφερθώ σε κάποιες παραγράφους εκθέσεως όπου αναφέρεται παραδείγματι ότι η γυναίκα στην πράσινη οικονομία στα κράτη-μέλη εργάζεται κυρίως μέσα στην οικογένεια αλλά λησμονεί ο εισηγητής την αλληλεγγύη μεταξύ των γενναιών και την γύρανση του πληθυσμού. Η πράσινη οικονομία δεν μπορεί χωρίς φιλελεύθερη ε, οικονομία να λειτουργήσει ικανοποιητικά. Θα επενθυμίσω τα όσα ίσχυαν στις χώρες μας στο παρελθόν και τα λόγια που ακούγαμε για την παρουσία της γυναίκας ε, στη γεωργία και την ε, μέρημνα για την οικογένεια. Εμείς την οικογένεια τη βλέπουμε ως ένα σύνολο και όχι ως ε, επιμέρους άτομα. Κοστέλο. Κοστέλο παρακαλώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλωσορίζω την ε, έκθεση και συγχαίρω τον εισηγητή. Είναι πολύ σημαντική η ενσωμάτωση της διάσταση του φύλου και όταν συζητούμε τα θέματα του περιβάλλοντος οι γυναίκες ως εργαζόμενοι είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες ε, στην καινοτομία και στην αναζωογόνηση αλλά κυρίως στην καινοτομία και την ε, δημιουργική οικονομία και πρέπει να ζητήσουμε και για τις γυναίκες τη θέση που τους αρμόζει σε μια πιο πράσινη οικονομία. Πρέπει να είναι παρούσες και στα όργανα λήψη αποφάσεων, να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον, για τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία, για να ενισχύσουν την ισότητα και τη δημοκρατία. Ιδιαίτερα στι αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η πρόσβαση στο είδωρ ή η αξιοποίηση της βιομάζας για, λόγους, ε, για ανάκτηση ενέργειας, είναι πολύ μεγάλη σημασία ε, και πρέπει να συμπεριλάβουν και τι γυναίκε. Πρέπει λοιπόν να δοθούν οι κατάλληλες στην πράσινη οικονομία. Ιδιαίτερα θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη για επενδύσεις και στα μέσα μας των συγκοινωνιών για ε, να λειτουργήσουν κατά τρόπον ενσωμάτωσης, κοινωνικής ενσωμάτωσης, όχι αποκλεισμού δηλαδή, αλλά και πράσινης οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπένοβα, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η πράσινη οικονομία μπορεί να χαρακτηριστεί οικονομία αηφορίας και βλέπουμε ότι όχι μόνο οι οικονομικές δραστηριότητες αλλά και η κοινωνική αηφορία αναφέρεται και πρέπει να είναι σεβαστή. Όλες αυτές τις διαφορετικές πτυχές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το φύλλο, την ε, θρησκεία, την ε, οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των ατόμων. Μια και η ρόλη των φύλων είναι διαφορετική, η συμμετοχή των γυναικών και η επίπτωση των γυναικών είναι διαφορετική από ό,τι σε σχέση με τους άνδρες. Υπάρχει δυστυχώς η αρνητική διακριτική μεταχείριση. Αυτή η ανισότητα μεταξύ μεταξύ των φύλων συνιστά, αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Η επιδίνωση ε, των όρων σε σχέση με το περιβάλλον έχει άμεσες επιπτώσεις στις ίδιες τις γυναίκες και τις πιο φτωχές γυναίκες. Το 70% είναι ε, όσον αφορά τους φτωχούς ε, γυναίκες. Οι γυναίκες δεν εκπροσωπούνται επαρκώς ούτε και όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το περιβάλλον, για τα θέματα τα δημοσιονομικά, τον προϋπολογισμό κτλ. Η κυρία Ρόμεβα παρακαλώ. Κύριε Στρομέβα, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Γκούσταυσον και για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε σε σχέση με την εκπόνηση της εκθεσής του. Είναι γεγονός ότι η απουσία ε, στις συνιστώσεις του φίλου αυξάνει την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το είδαμε αυτό. Γι' αυτό η ένταξη της πτυχής του φίλου και η αντιμετώπιση της ανισότητας ε, συνιστά σημαντική υπόθεση. Αυτό είναι εκείνο οποίο θέλουμε να ληφθεί υπόψη στην έκθεση και εκτιμούμε ιδιαίτερα ότι έχουμε και δύο τροπολογίες που καταθέσαμε που λαμβάνονται υπόψη. Τον εξειδικευμένο ρόλο τον οποίο έχουν οι γυναίκες σε σχέση με την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκθέσεις είναι γεγονός ότι οι γυναίκες πλήττονται πολύ περισσότερο λόγω της κρίσης ε, σε σχέση με τους άντρες ε, πολύ περισσότερο από αυτούς και σε μια τέτοια ε, η οικονομία πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη. Είναι μια ευκαιρία να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης λοιπόν προς όφελο των γυναικών. Ευχαριστώ. Η κυρία Τικάου παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οι κλιματικές αλλαγές ε, και η απώλεια βιοπικιλότητας απειλούν ε, την ε, κοινωνική ευημερία και την διαβίωση των πληθυσμών μας. Ζητώ από τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα υπέρ των γυναικών για να μπορέσουν να βοηθήσουν ώστε οι γυναίκες να συγκλίνουν στην οικογενειακή ζωή και επαγγελματική ζωή και την εισαγωγή καινοτομιών ιδιαίτερα ιδιαίτερα όσον αφορά την οικολογία και τις ε, υπηρεσίες. Θέλουμε να υποστηριχθούν οι γυναίκες για τις μικροπιστώσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά μικροεπιχειρήσεις όπου θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν και θα μπορούσαν μέχρι 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης να δημιουργηθούν. Γι' αυτό ζητούμε από τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν μαθήματα κατάρτισης ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών σε αυτές τις νέες τεχνολογίες και τις αναδυόμενες τεχνολογίες που έχουν σημασία σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ζητούμε να υιοθετήσουν πολιτικές φορολογικές τα κράτη-μέλη που θα μπορούν να έχουν θετικές επιπτώσεις για τις επενδύσεις και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τσίσκοβα παρακαλώ, τελευταία που θα λάβει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αρχικά Ήθελα να ομιλήσω για την επόμενη έκθεση. Παρόλα αυτά όμως κάποιες ε, παρεμβάσεις που έγιναν θα μπορούσα να τις ε, σχολιάσω. Εκτιμώ ιδιαίτερα τους συναδέλφους αλλά οι παρεμβάσεις αυτές ε, με οδήγησαν και εγώ να θελήσω να σχολιάσω αυτά τα θέματα. Άσχετα αν πρόκειται για γυναίκες ή άνδρες στον ρόλο της πράσινης οικονομίας πρέπει όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να δράσουν. και γι' αυτό είναι αναγκαίο η ισότητα να υποστηριχθεί ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες και πρέπει αυτή να είναι η σημερινή πολιτική που θα ισχύει ιδιαίτερα σε μια χρονική συγκυρία όπου οι γυναίκες έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά αλλά θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται και συνεχίζουν να εργάζονται για να μπορούν από κοινού με τους συζύγους τους να μεριμνούν για τα παιδιά και να ασχολούνται με τη γονεϊκή μέρημνα. Ακόμα και όταν εργάζονται στην γεωργία όπου η οικογένεια μπορεί να συνεργαστεί με θετικό τρόπο. Δεν μπορώ να συμφωνήσω να υφίστανται κυρώσεις στα παιδιά επειδή εργάζονται οι μητέρες τους. Θέλω να υποστηρίξω την ιδέα που τονίζεται από την έκθεση αυτή ώστε να έχουν δυνατότητες πολυμορφοποίησης απασχόλησής του οι γυναίκες. Uh, Mr. Ο κύριος Επίτροπος Νταλή θα λάβει τελευταίο τον λόγο παρακαλώ. Εξ ονόματο της Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον κύριο Γκούσταυσεν για την έκθεσή του. Να ευχαριστήσω επίσης και την Επιτροπή Γυναικών και ισότητα των φίλων για την παρέμβασή της. Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών και η προστασία των δικαιωμάτων τους είναι κάτι που συνδυάζεται με την αηφόρο ανάπτυξη και με την πρόοδο στον τομέα της πράσινης οικονομίας. Αυτό είναι απαραίτητο σε τομείς όπως η διατροφή, αηφόρος γεωργία, προστασία των υδάτων κτλ. Η συζήτηση αυτή είναι ιδιαίτερο εύθετη επίσης ε, στα πλαίσια των στόχων που έχουμε θέσει, όπου το θέμα των φύλων παίζει σημαντικό ρόλο. Η Agenda Plus 20 έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις και έχει προκαλέσει ενδιαφέρον μεγαλύτερο ίσως από ό,τι περιμέναμε και στον τομέα της ισότητας των φύλων. Η ενίσχυση λοιπόν της θέσης της γυναίκας είναι κάτι πέραν από τις θέσεις που είχαν αποφασιστεί στο ε, Johannesburg και προσπαθούμε να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε τα πολιτικά μας οράματα να τα κάνουμε πραγματικότητα στα πλαίσια της ισορροπίας των φύλων και της ενίσχυσης της θέσης της γυναίκας σε πάρα πολλούς τομείς. Να συγκεντρώσω την προσοχή μου σε ένα άλλο θετικό θέμα που πολλές φορές αγνοείται σε σχέση με το Ρίο Το λεγόμενο mainstreaming σε πάρα πολλά κεφάλαια των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν σχέση και με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της θέσης των γυναικών, της καταπολέμησης της ένδυας. Στο Ρίο υπήρξε συμφωνία για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών σε, στην Ήπεθρο ιδιαίτερα και κυρίως σε σχέση με την παραγωγή τροφίμων δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους μικρούς παραγωγούς και κυρίως τις γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε μικροδάνεια, σε κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, ε, κατάρτιση και τεχνολογία. Η εισαγωγή της διάστασης του φύλου στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε όλες αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα βοηθήσει πολύ το Ρίο αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Οι προσπάθειες που γίνονται για την μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς αποκλεισμούς και σε μια πράσινη οικονομία τώρα έχει ξεκινήσει ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή και αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα τεκμηριώνονται σωστά στο παρόν κείμενο. Θα ελπίζουμε σε μια καλύτερη στο μέλλον συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Αρμόδια Επιτροπή. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Η συζήτηση τελείωσε. Η ψηφοφορία ε, θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Σα ευχαριστώ. Το επόμενο σημείο στη ημερήσια διάταξη είναι τώρα η έκθεση τη ε, κυρία Γκαρσία Πέρετ Συνθήκε εργασία των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών». Θα λάβει τον λόγο η κυρία εισηγήτρια. Τέσσερα λεπτά παρακαλώ κυρία Πέρετ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο τομέα των υπηρεσιών είναι περίπου το 70% τη συνολική απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 83% της, ε, του